Uh, uh, Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο δεύτερο μέρος της συνεδριάσεώς μας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς για σήμερα. Ήταν πολύ άσχολο το πρωινό μας, καλύψαμε πολλά σημεία, προχωρήσαμε αρκετά στον αφορά τους συμβιβασμούς. Αυτό ήταν μια καλή εισαγωγή στην απογευματινή συνεδρίαση με την Ελληνική Προεδρία και με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Κώστα Χατζηδάκη στη συνεδρίασή μας. Δεν του λέω καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πέρασε ήδη πολύ καιρό εδώ. Ε, το γνωρίζουμε όλοι. Κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Καταρχήν, καλωσορίζω πάντα το ακροατήριο από το διαδίκτυο, διότι εκπέμπουμε στο διαδίκτυο. Ε, είναι πολύ καλό να ξέρει κανείς ότι πολλοί ακούν το διαδίκτυο. Έχουμε ένα, μια νέα εφημερίδα την μπορεί να διαβάσετε και στο διαδίκτυο και καλωσορίζω τους συναδέλφους. Έχουμε και φοιτητέ ε, από το Πανεπιστήμιο του Άστον στο Μπέρμιχαμ, όπου εκεί είμαι επίτιμος καθηγητής επιστημών, ε, φυσικών επιστημών και τους καλωσορίζω. Όπως, ε, όπως είπα, ο Κώστας δεν χρειάζεται παρουσίαση και σύσταση σε πολλούς από εμάς. Κώστα ήσουν διεκεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, επιφανές και δραστήριο μέλος του ΕΛΚ στη θητεία του στο Κοινοβούλιο. Τον ξέραμε πολύ. Με τα χαρά σας συναντήσαμε τον Αύγουστο που ήρθαμε την προσωπία μελών. Πολλοί από αυτούς είναι εδώ σήμερα. Όταν μας μίλησες για τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και κάποιες από τις φιλοδοξίες σου για την Προεδρία, είναι πολύ καλό, υπέροχο που είσαι εδώ μαζί μας για να μας μιλήσεις για το ρόλο σου, πολύ κρίσιμο ρόλο του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και έχεις και πάρα πολλές άλλες ευθύνες στο χαρτοφυλάκιό σου, στην ελληνική κυβέρνηση. Ενδιαφερόμαστε πολύ να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις και οι συνάδελφοι θα σου ετοιμάσουν ερωτήσεις για την πρόοδο διαφόρων χαρτοφυλακίων. Έχω ήδη έναν κατάλογο ομιλητών. Λοιπόν, θα ακούσεις τα ονόματα μετά. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσω τον πρώτο γύρο στους συντονιστές για να υποβάλουν ερωτήσεις όπως συνήθως και μετά θα πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι. Μεγάλη μου χαρά ε, να σου δώσω το μικρόφωνο να μας μιλήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Μάλκο. Πραγματικά είναι χαρά για μένα να είμαι εδώ και θα έλεγα είναι και συγκινητικό για μένα διότι ήμουν μέλος αυτού του κοινοβουλίου για 13 χρόνια. Από το 1994 μέχρι το 2007 δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για να προεδρεύοντα του Συμβουλίου να είναι επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν είναι θετικό για το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει αυτά έχει ζωή. Επίσης Πρέπει να σας θυμίσω ότι ήμουν και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για δυόμιση χρόνια, της Επιτροπής αυτής. Ασχολήθηκα λοιπόν με τα θέματα που αντιμετωπίζετε τώρα και τα αντιμετώπισα εδώ και κάποια χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Μάλκολμ ήταν ο συντονιστής μου. Και θα προσπαθήσουμε να είμαστε συντονισμένοι ακόμα και τώρα και να έχουμε συντονισμένες δράσεις. Όμως, ξέρετε, η ελληνική προεδρία είναι αρκετά ιδιαίτερη προεδρία, διότι διαρκεί μόνο ένα τρίμηνο. Και είναι μπροστοβαρής προεδρία, πρέπει να κινηθούμε τάχιστα και να πετύχουμε αποτελέσματα. Η προεδρία για μας είναι μια πραγματική πρόκληση, διπλή πρόκληση θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα διότι συμπίπτει με τις ευρωεκλογές. Είναι κρίσιμη η περίοδος αυτή. Πρέπει να ολοκληρώσουμε κάποια θέματα, θα πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα και να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, έχουν πραγματικά προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα η ελληνική προεδρία είναι σημαντική όσον αφορά την Ελλάδα, τη χώρα την ίδια, την Ελλάδα, διότι είναι μια δυνατότητα, ίσως είναι μια ευκαιρία για μας να διορθώσουμε τις ζημίες που έχουν προκληθεί στην εικόνα της χώρας κατά τα τελευταία χρόνια. Απότερος σκοπός θα έλεγα είναι να σε εκπλήξουμε θετικά. Πώς? Έχοντας μια πραγματιστική ατζέντα, χωρίς να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, εστιαζόμενοι επί συγκεκριμένων ζητημάτων, επί νομοθετικών χαρτοφυλακίων και ξέρετε πιστεύουμε ότι αν έχουμε μια πραγματιστική προσέγγιση, αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάποιους συμβιβασμούς μαζί σας, αυτό σίγουρα θα είναι καλό για την ελληνική προεδρία, αλλά και για το Κοινοβούλιο και πάνω απ' όλα για την Ευρώπη και για τους πολίτες της. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δράσουμε και βέβαια είναι αυταπόδεικτο και αυτονόητο, αλλά πρέπει να το επαναλάβω. Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο, με αυτή την Επιτροπή όλος ιδιαίτερος, με τον Προέδρο, τους συντονιστές και βέβαια τους εισηγητές και όλα τα άλλα μέλη, ούτως ώστε να έχουμε Επιτυχής τριμερής διαλόγους, ούτως ώστε να δώσουμε αποτελέσματα, να πετύχουμε αποτελέσματα. Έτσι θα εργαστούμε και στο τέλος πιστεύω ότι θα είμαστε επιτυχείς, διότι είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε όλοι μας. Έρχομαι τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Θα ήθελα να πω ότι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, του οποίου θα προεδρεύω επί το επόμενο εξάμεινο, η δουλειά μας πρέπει να αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να βελτιώσουμε επίσης την ανταγωνιστικότητα προστατεύοντας τους καταναλωτές. Η ανταγωνιστικότητα είναι κλειδί για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και για να καταπολεμήσουμε την αυξανόμενη ανεργία Έχουμε δραματική εμπειρία αυτού στην Ελλάδα, αλλά και είναι μια ενεργεία που αντιμετωπίζει στο σύνολό της η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς είναι ένα απαραίτητο βήμα, ώστε να δώσουμε μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και να ξαναμπούν στον δρόμο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ελληνική προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων που είναι η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης, να προωθήσουμε την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη, καθώς και να βελτιώσουμε το πλαίσιο για τους καταναλωτές και το νομικό πλαίσιο. Αυτές θα είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της Προεδρίας. Επιτρέψτε μου τώρα, μετά από αυτή τη γενική περιγραφή των προτεραιοτήτων μας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ακροθυγώς στους στις βασικές νομοθετικές μας ε, προτεραιότητες, οι οποίες μετρούν περισσότερο στο τέλος και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της δικής σας επιτροπής, δηλαδή η τεχνική εναρμόνιση και τα συναφή ζητήματα, τα πακέτα ταξιδίων, η ασφάλεια των προϊόντων και η υποπτία της αγοράς και τα σχετικά πακέτα, και πρόταση οδηγίας για ηλεκτρονικά τιμολόγια στις δημόσιες προμήθειες και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ακριβής μπορώ ως Προεδρεύων. Εσείς έχετε το πλεονέκτημα να μιλάτε, να συζητάτε με διαφορετικό τρόπο, να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία από ότι εγώ σε αυτή τη φάση. Καταρχάς, παρόλο που πιστεύω ότι είναι, δεν είναι το πιο δημοφιλές θέμα στο πρόγραμμά σας, ούτε και το πιο εύληπτο για τους πολίτες, θέλω να εκφράσω μεγάλη ικανοποίηση. Για την προσωρινή συμφωνία που πετέχθη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την οδηγία για τον νέο εξοπλισμό, ραδιοφωνικό εξοπλισμό, ξέρω ότι η συγγήτριά σας ήταν η κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς αυτήν προσωπικά. Είναι το πρώτο χαρτοφυλάκιο που ολοκληρώνεται επί ελληνικής προεδρίας όσον αφορά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και γι' αυτό έπρεπε να κάνω ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό, κυρία Βάιλερ. Την ξέρω το 1994, έτσι δεν είναι, ήμασταν μαζί. Στην Επιτροπή Απασχόλησης τότε. Α, κοινωνικών υποθέσεων. Εξωσημείωτη η δουλειά που έκανε η Ιρλανδική και η Λιθουανική Προεδρία ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Προεδρία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι δε περαιτέρω η συμβαστική μας πρόταση για τον εξοπλισμό που λειτουργεί υποπίεση, η κυρία Ρόιτοβα είναι η συγγήτρια είναι κάτι που συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 1 για να δοθεί διαπραγματευτική εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την μεταφορά της καταχώρησης οχημάτων, μερική εντολή δόθηκε στον κύριο Μάντερς 18 18 Δεκεμβρίου και τώρα προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας με τον εισηγητή σας και την επιτροπή σας για να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό συμφωνία για την έγκριση της εν λόγω πράξης πριν το τέλος της θητείας. Για να πω την αλήθεια, δεν είμαι ο υπεύθυνο υπουργό για αυτό το θέμα, αλλά το Υπουργείο Μεταφορών ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, αλλά πρέπει να αναφερθώ στο θέμα αυτό, διότι είναι σημαντικό θα έλεγα για εσά και για μας και πρέπει να εξετάσουμε επίσης, να ξεκινήσουμε την εξέταση του άλλου ζητήματος της οδηγίας ε, για τις ε, ηλεκτρονικές κλήσεις. Μου είπαν ότι η συγγήτριά σας είναι η κυρία Σαρδάνοβα για το e-call. Είστε εδώ. Ευχαριστώ που είστε παρούσα. Μόλις ξεκινήσαμε, δεν ξέρω πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε, εξαρτάται και από τους δυο μας αυτό και θα δούμε. Τούτων λεχθέντων, όσον αφορά την τεχνική εναρμόνιση, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την οδηγία για τα ταξίδια. Παρόλο που το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας ασχολείται με το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με το ζήτημα, διότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες της δικής σας Επιτροπής. Ο κύριος Μάγιο ο εισηγητής, δεν είναι εδώ ακόμα. Είναι παλιός φίλος. Η ελληνική προεδρία δίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση οδηγίας. Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για μας. Προφανές είναι αυτό. Στα τέσσερα συνεδριάσεις ομάδας εργασίας που έλαβαν χώρα επί Λιθουανικής Προεδρίας, 11 από τα 29 άρθρα ε, συζητήθηκαν και εξετάστηκαν. Η Ελληνική Προεδρία έχει σαν στόχο να διεκπαιρεώσει την πρώτη ανάγνωση και να ετοιμάσει έκθεση προόδου για την επικείμενη Ιταλική Προεδρία. Θα θέλαμε να διεκπαιρεωθεί το θέμα αυτό, αλλά δεν εξαρτάται από εμά. Εξαρτάται από την επιτευχθήσα ή μη επιτευχθήσα πρόοδο, εξαρτάται από άλλα κράτη-μέλη και θέλω να είμαι ειλικρινή. Αυτό είναι ο στόχο μας και ελπίζω να είμαστε επιτυχείς η ηλεκτρονική τιμολόγηση στους διαγωνισμούς στις κρατικές προμήθειες και η ασφάλεια των προϊόντων και η υποπτία της αγοράς και τα διάφορα αυτά σχετικά πακέτα είναι βασικές δράσεις στην ενιαία πράξη, ε, την πράξη για την ενιαία αγορά υπαριθμών 2 και έχουν ε, ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική προεδρία. Θα ξεκινήσω από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι πιο ευχάριστο θέμα. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, να συγχαρώ την κυρία Κολιν Λάγκεν. Έξοχη η δουλειά, το αποτέλεσμα που πέτυχε στις ψηφοφορίες, είχε ομόφωνη υποστήριξη ε, η έκθεσή της από την Επιτροπή σας στις 17 Δεκεμβρίου. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει πάρα πολύ υψηλή οικονομική σημασία και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες οικονομίες Θέλω να μοιραστώ μαζί σας την πεποίθηση ότι μπορούμε μαζί να πετύχουμε σε πρώτη ανάγνωση συμφωνία και προώθηση αυτού του θέματος επί ελληνικής προεδρίας. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί ε, στις 14 Ιανουαρίου και ο χθεσινός τριμερής διάλογος κατέληξε στο να εκρεμεί ακόμα μόνο η προθεσμία όσον αφορά την ε, ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας. Πρόεδρε, κύριε Χάρμπουρ, θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας για να ξεπεράσουμε τα εναπομένοντα εμπόδια, ώστε να έχω μια συμφωνία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, ένα την Παρασκευή. Παρασκευή. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσετε. Στο κάτω-κάτω έχουμε κοινού στόχους όσον αφορά το θέμα αυτό. Μετά πρέπει να κλείσω τα σχόλιά μου αναφερόμενος σε άλλο επίμαχο ζήτημα, σημαντικό, την ασφάλεια των προϊόντων και το πακέτο για την εποπτεία της αγοράς παρά την επικοδομητική δουλειά των εισηγητών σας, της εισηγήτριάς σας, της κυρίας Σάλντερ Μόζε και της κυρίας Πιέτη Κάιναν, οι εξελίξεις υπήρξαν λιγότερο θετικές όσον αφορά το πακέτο για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε το προβληματικό άρθρο 7 του κανονισμού για την ασφάλεια των προϊόντων όσον αφορά τη ρήτρα για το που είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα, made in, και υπάρχει διαίρεση μεταξύ κρατών μελών στην Κορεπέρα 1. Δεν αποτελεί μυστικό, γνωρίζετε τις ε, λεπτομέρειες δεν θα έπρεπε να αναφερθώ σε συγκεκριμένες ε, πτυχές των διαφορών. Η Προεδρία πρέπει να δράσει ως καταλήτης, να είναι επικοδομητική και πιστέψτε με, η Ελληνική Προεδρία έχει υποβάλει επικοδομητικές συμβαστικές ε, προτάσεις για να ξεπεραστεί η αποτελμάτωση διαπραγματεύσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές για να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών επ' αυτού. Γι' αυτό δεν παρετούμεθα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε παρά τις δυσκολίες. Αυτό είπα και στην ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία στον πρεσβευτή μας που ασχολείται με το θέμα αυτό Βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα ότι έχετε χρονική πίεση λόγω των εκλογών. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, να βρουν τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, έναν κοινό παρανομαστή μάλλον. Είναι δύσκολο, δεν υποτιμώ τις ε, δυσκολίες, όμως θα θέλαμε να το σώσουμε το πακέτο στο βαθμό του δυνατού, όσο μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κάποιες εναλλακτικέ, ας πούμε κάποιες ευφυείς λύσεις, ό,τι είναι δυνατόν, ε, ούτω ώστε να πετύχουμε συμφωνία πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, διότι η εναλλακτική θα είναι να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Η εναλλακτική είναι να έχουμε νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέα πρόταση, νέο κοινοβούλιο, νέα συζήτηση. Το νωρίτερο συμφωνία μπορούμε να πετύχουμε τέλος του 2015 πιθανότατα. Αυτό δεν είναι καλό για την Ευρώπη, δεν είναι καλό για την εσωτερική αγορά, δεν είναι καλό για τους καταναλωτές. Γι' αυτό εξακολουθούμε τις προσπάθειές μας. Βέβαια δεν τρέφουμε αυτά πάτες, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβούν θαύματα σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, ναι. Εν πάση περιπτώσει δοθέντος ότι έχουμε κάποιο χρόνο, κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το χρονικό αυτό διάστημα, ούτως ώστε να έχουμε πιθανότατα κάποια αποτελέσματα. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Προσπάθησα να είμαι ακριβής. Αν λησμόνισα κάτι μπορούμε να το συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαι στη διάθεσή σας Είμαι εδώ να ακούσω τις απόψεις σας και πάνω απ' όλα είμαι εδώ για να συνεργαστώ μαζί σας. Δεν ξέχασα ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι εδώ, ήμουν παλιό συνάδελφό σας, ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι εδώ στο κοινοβούλιο και πιστέψτε με, ειλικρινά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Βέβαια για την Ελληνική Προεδρία αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Κώστα που μας είπες ακριβώς το, ποιο είναι το πρόγραμμά σας. καλό ξεκίνημα, έχεις δίκιο και ελπίζω ότι αν πετύχουμε συμφωνία αυτή την εβδομάδα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα έχουμε ολοκληρώσει δύο χαρτοφυλάκια. Οπότε ξεκινάμε καλά. Καλό τους συντονιστές να υποβάλουν ερωτήσεις. Ένας-ένας μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μέχρι τις μισή χρόνο, έτσι δεν είναι. Ο κ. Σβάπη, η κυρία Κέπχαρτ, ο κ. Μάντερς και η κυρία Ρούλε. Ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ μου Κώστα, κύριε Υπουργέ, θερμό καλωσόρισμα σου εύχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς σε σκεφτόμαστε, όπως είπες και εσύ ότι άφησες ένα κομμάτι της καρδιάς σου εδώ και χαίρομαι ε, που θα σε βλέπουμε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, στην οποία ευχόμαστε καλά αποτελέσματα. Ένα θέμα που αναφέρθηκε ήδη είναι οι ηλεκτρονικές τιμολογήσεις. Εκεί ε, θα χρειαστεί ευελιξία από το Συμβούλιο θα έλεγα εγώ. Το θέμα είναι αν για το εθνικό επίπεδο έχουμε, ε, αν θα βρούμε 18 με 24 μήνες συμβιβαστική λύση στο Συμβούλιο. Ε, καλό θα ήταν το ο φάκελος της κυρίας Κρόνιν Λάγκεν να ε, κολλήσει στην προθεσμία 18-24 μήνες για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Για την υποεθνική παραμένει το, η προθεσμία των 30 μηνών. Παρακαλώ κατεπηγόντως να προλάβουμε και να καταφέρουμε την Παρασκευή να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση όταν θα συνέλθει πάλι η ομάδα του Συμβουλίου. Δεύτερον, ε, δεν αναφέρθηκε, ε, ίσως ε, ο Υπουργός Μεταφορών θα είναι υπεύθυνος, θα πρέπει να δούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Και στην Γερμανία και από αλλού μάθαμε ότι 16 εκατομμύρια email accounts έπεσαν θύματα hackers και είναι πολύ σημαντικό και για την προστασία των δεδομένων ε, όσο πιο γρήγορα σε, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να δώσουμε μια απάντηση και να φροντίσουμε ούτω ώστε οι αρμόδιοι πάροχοι να επενδύσουν περισσότερο στην αντοχή των συστημάτων τους, στην ε, και θα ήθελα να ξέρω τι ατζέντα έχει η ελληνική προεδρία σε σχέση με την ενημέρωση και την οδηγία για να έχουμε ταχύτατα αποτελέσματα. Η Επιτροπή αύριο Πέμπτη θα ψηφίσει και από ό,τι κατάλαβα ο συνάδελφος Γκαρσία Ραμμόν από τους σοσιαλιστές δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή αλλά νομίζω ότι βρήκαμε καλές συμβιβαστικέ λύσεις και θα ψηφίσουμε σχεδόν ομόφωνα οπότε θα μπορούσαμε γρήγορα να βρούμε μια λύση. Ε, κυρία, δεν θέλω βέβαια να προδικάσω αυτά που θα πούν οι κυρίες Σάλντε Μόζερ και ποιετικά είναι, αλλά θέλω να πω ότι όλα τα άλλα άρθρα που δεν είναι επίμαχα στο πακέτο για την ασφάλεια θα έπρεπε να τα κατοχυρώσουμε από αυτό το κοινοβούλιο γιατί είναι κρίμα να χαθούν. Ευχαριστώ. Ωραία, ένα-ένα. Ανδρέας για το, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια κάναμε το καλύτερο δυνατό για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Ε, είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, πιστεύω. Πρέπει να συζητήσουμε και κάποια, με, κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε στο μυαλό μας κάποιες ιδέες που ίσως αποβούν επικοδομητικές για να ε, επιτύχουμε το στόχο μας αυτόν και χρειάζεται κάποια ευελιξία και από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο όμως. Τέλος πάντων, στο παρελθόν όλοι μας καταφέρναμε να λύνουμε ακόμα και πιο δύσκολα προβλήματα από αυτό. Κατανοώ την ανάγκη για γρήγορη μεταφορά στο εθνικό επίπεδο της οδηγίας για προφανείς λόγους. Καταλαβαίνω και τις δυσκολίες ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες εθνικές ευαισθησίες. κάνουν ό,τι μπορούμε. Τώρα, για το δεύτερο θέμα, δηλαδή την ασφάλεια των πληροφοριών, ο Μάλκολ μου είπε ότι εσύ είσαι ο εισηγητής, το ξέρεις εσύ το θέμα, εγώ όχι. Για τον απλό λόγο ότι δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να μεταφέρω το μήνυμά σου στον Υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, ο οποίος το χειρίζεται το θέμα, ώστε να απαντηθεί η ερώτησή σου. Τη σημειώνουμε. Αλλά οι πολιτικοί πρέπει να λένε την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ την αλήθεια λέω, δεν το ξέρω το φάκελο, γιατί δεν το εγχειρίζομαι εγώ. Η Εύελιν Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω εδώ. Και ως εισαγωγική παρατήρηση θέλω να πω ότι σίγουρα ε, ήταν καλό που υπήρξατε Ευρωβουλευτής, γιατί εμείς ξέρουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, διότι άλλοι υπουργοί ε, μας έδωσαν διαφορετική εικόνα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπουμε πρώην συναδέλφους που, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί. Αναφέρατε ένα θέμα στην ομιλία σας που μας ενδιαφέρει εμάς πολύ τους ε, σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή και δημιουργούν και τις περισσότερες θέσεις εργασίας στα κράτη μας και στην Ελλάδα, την Ισπανία και άλλες χώρες ε, η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει τεράστια σημασία και οπωσδήποτε θα πρέπει αυτό να είναι μια πολιτική προτεραιότητα όπως και το θέμα της αναβιομηχάνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ε, λογικό και σωστό τρόπο. Θέλω να απευθύνω και μία έκκληση ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό για τους πολίτες είναι ένα θέμα εξόχως σημαντικό. Θέλω να σας υποστηρίξω στις προσπάθειές σας για να φροντίσετε ότι ο φάκελος αυτός θα προχωρήσει το ταχύτερο και το καλύτερο δυνατόν. Γιατί οι πολίτες θέλουν ασφάλεια, θέλουν ασφαλή προϊόντα, θέλουν όμως και ενημέρωση, πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων. Βεβαίως υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και εδώ στο Κοινοβούλιο, όμως καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση που είναι και η εντολή, αν θέλετε, του Κοινοβουλίου. Και σας καλώ να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν και στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να υπάρξει αυτή η σύμφωνη γνώμη. Και η έκκληση αυτή δεν είναι προσωπική προς εσάς αυτή, αλλά προς το Συμβούλιο συνολικά, η έκκληση είναι η εξή. Στι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταργήσει την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αλλά το Συμβούλιο εξακολουθεί να εργάζεται με βάση την αρχή τη ομοφωνία. Και αυτό πολύ συχνά παρεμποδίζει την πολιτική, την άσκηση τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως βοηθήσετε και εδώ αυτό το λάθος που γίνεται στο Συμβούλιο να αποκατασταθεί, ούτως ώστε να είναι ευχερέστερη η διαμόρφωση της πολιτικής. Ε, πριν φτάσω στο τελευταίο για το οποίο γελάει ο πρόεδρος, θα μιλήσω λίγο, είναι πιο ευχάριστο για μένα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. λοιπόν, ε, είναι προτεραιότητά μας δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του επόμενους τρεις μήνες, αλλά υπάρχει ένα μείζον θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την ώρα στην Ευρώπη, ιδίως στις χώρες που πλήττονται από την κρίση που έχει να κάνει με το access to finance, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Οι δικέ μα επιχειρήσει δανείζονται στην Ελλάδα με επιτόκιο 19, 10%, 9%. και, και πραγματικά διαρωτώ με πολλέ φορέ και τι είδου εσωτερική αγορά είναι αυτή και τι είδου ανταγωνισμό υπάρχει όταν άλλε επιχειρήσει αλλού δανείζονται με 3% και με 4% και με 5%. Είναι ένα πρόβλημα και εκεί έχει συζητηθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχει δοθεί εντολή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παρουσιάσει καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία και προϊόντα. Θα δούμε μέχρι στιγμή οι αντιδράσει των περισσότερων κρατών μελών σε σχέση με τι ιδέε που προτάθηκαν δεν είναι θετικέ. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά το θέμα τη ρευστότητα, το θέμα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ειδικά για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι πολύ σημαντικό. Όπω σημαντικό είναι για μα και το θέμα τη βιομηχανική πολιτική συνολικά, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπω η γραφειοκρατία, πρέπει να τονιστεί και να τονωθεί η διάσταση της ε, ε, καινοτομίας, του innovation και επίσης πρέπει να δούμε επιτέλους στην Ευρώπη το θέμα του κόστους της ενέργειας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τόσο καιρό μιλάγαμε και σωστά κάναμε για το περιβάλλον ε, και πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για το περιβάλλον, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά χωρίς βιομηχανία η ανεργία θα αυξηθεί. Η στήριξη της βιομηχανίας είναι στην πραγματικότητα κοινωνική πολιτική. Και αυτό είναι που πρέπει να κατανοηθεί από αυτούς που ξεχωρίζουν τα δύο πράγματα μεταξύ τους, πιστεύοντας ότι μπορεί να υπάρξουν επενδύσεις χωρίς επενδυτές και ανάπτυξη χωρίς βιομηχανία. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τώρα έρχομαι στο πιο δύσκολο, ε, στο Product Safety Package. Ξέρω ότι έχετε συμφωνήσει. Ξέρω ότι και σε εσά υπήρξαν συζητήσεις και έχετε καταλήξει σε ένα κοινό παρανομαστή. Έχουμε ήδη κάνει προτάσεις. Οι προτάσεις οι οποίες έχουμε κάνει και, και, είναι διαφορετικές προτάσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Τρεις εναλλακτικές προτάσεις καταθέσαμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν προχώρησαν. Ε, σήμερα κατατέθηκε και άλλη πρόταση, ε, η οποία και αυτή δεν προχώρησε. Ε, και, και όπως σας είπα η εντολή μας στον αρμόδιο Έλληνα πρέσβη που το χειρίζεται αυτό είναι να συνεχίσει να διαπραγματεύεται. Ε, όποια ιδέα έχετε όπως είπα και πριν που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το θέμα στη διάθεσή σας είμαστε. Και αυτό ισχύει σε δύο επίπεδα. Πρώτον στο επίπεδο της ουσίας μήπως υπάρχει καμιά ιδέα που μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει για να ξεπεράσουμε το deadlock, το, το αδιέξοδο. Και το, και το δεύτερο α, είναι στο διαδικαστικό επίπεδο. να δούμε πώς από πλευράς διαδικασίας, από πλευράς χειρισμών κτλ. Ποια θα ήταν η κίνηση εκείνη, οι κινήσεις εκείνες που ε, μπορεί να μας βοηθήσουν. Προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ την επόμενη Δευτέρα για άλλους λόγους στις Βρυξέλλες. Αλλά θα είμαι εδώ. Ε, και νομίζω και την Τρίτη το πρωί. Εάν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας με τους συζητητές, με εσά, με όλους, να καθίσουμε και προσωπικά να συζητήσουμε, να δούμε αν μπορεί κάτι να γίνει. Αλλά επίσης ο πρέσβης, ο κ. Παπασταύρου, ε, είναι συνέχεια εδώ και ε, έχει σαφή κατεύθυνση να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο προκειμένου να, να βρούμε κάποια λύση. Ξέρετε, δεν είμαστε ταχυδακτηλουργοί. Δεν είμαστε μάγοι, δεν μπορούμε να, να, να βρούμε λύσεις όταν υπάρχει μια κάθετη άρνηση από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Ε, ε εμείς πρώτοι από όλους θέλουμε να υπάρξει αποτέλεσμα διότι μας ενδιαφέρει να κλείσουμε αυτό το ντοσιέ. Είναι, είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει τέσσερις εναλλακτικέ προτάσεις μέσα σε δύο εβδομάδες. Ε, αλλά από εκεί και πέρα ε, και η φαντασία εξαντλείται. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω και, και, γι' αυτό είμαστε στη διάθεσή σας για να δούμε πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα, τα ζητήματα αυτά, τα προβλήματα. Well, thank you, thank you very much. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε σήμερα το βράδυ μια σχετική συνεδρία. Θα το συζητήσουμε βεβαίω. Ο κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε πρώην συνάδελφο να είναι τώρα η υπουργό και να συνεργαζόμαστε μαζί του. Αναφερθήκατε ε, στην ταξινόμηση των ε, αυτοκινήτων. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ε, συζητήσει πολλές φορές. Θες είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με το Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύση αν τα καταφέρουμε εντός των ε, χρονικών ορίων μας. Υπάρχει πάντα ε, χρονική πίεση σε αυτά τα θέματα. Ελπίζω όμως, ελπίζω, είμαι πεπισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Αυτό που θα ήθελα να σας πω και ε, ως πρώην Ευρωβουλευτής γνωρίζετε τι θα πει αυτό. Το Συμβούλιο συχνά έχει μια πολύ τεχνοκρατική προσέγγιση και στην πολιτική δεν, είναι μόνο, δεν υπάρχει μόνο νομοθεσία είναι μερικές φορές πρόκειται και περί του να δοθεί δυνατότητα στους πολιτικούς να δείξουν τι έχουν επιτύχει. Ελπίζω να μπορέσετε και εσείς να το μεταφέρετε αυτό ε, στην ε, ομάδα και στους συνεργάτες σας. Ε, κάτι που θα ήθελα να σας πω, μια και είστε προεδρεύων, έχουμε πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όλο και λιγότερη υποστήριξη υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να αρχίσουμε μεταρρύθμιση της ε, υπάρχουσας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε ελπίδα για το μέλλον, όπως κάναμε το 1957, όπως κάναμε το 1992 με την ε, έναρξη της εσωτερικής αγοράς. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο όνειρο για το πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς νομίζω με την ελληνική προεδρία μπορείτε να αποτελέσετε την αφετηρία. Ένα από τα βασικά προβλήματα κατά τα επόμενα δέκα έτη και το είπε και ο Ανδρέας Φαμπ, 590.000 άτομα χρειάζονται για το ίδιο ε, επίπεδο ευημερίας. Ε, ε, ελπίζουμε στην επόμενη επιτροπή να έχουμε έναν επίτροπο, αντί για πολυγλωσία, να έχουμε έναν επίτροπο γυράσκοντος πληθυσμού. Ευχαριστώ. <laughs> I have to explain. Να εξηγήσω. Πρέπει να φύγω από το κόμμα μου που είναι οι ε, φιλελεύθεροι. Είναι για τους ανθρώπους που είναι πάνω από 50. Αυτός είναι Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. No, what you said is... Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε κύριε Μάντερς. Ο ευρωσκεπτικισμός ε, είναι πραγματικός εχθρός ε, όχι μόνο για τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρώπης, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, για τους πολίτες της. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη Ευρώπη και πιο αποτελεσματική Ευρώπη. Και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας από την κρίση και πρέπει να ξανασκεφτούμε όσα κάναμε ως τώρα. Και για ποιο λόγο να μην ε, καταργήσουμε και πλεονάζουσα νομοθεσία, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, για να ε, υιοθετήσουμε μία πιο φιλελεύθερη προσέγγιση ε, σε σχέση με, την, με το μέλλον μας. Παράλληλα όμως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κάποιων διαρθρωτικών ε, κενών στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Χρειαζόμαστε ένα νέο ευρωπαϊκό όνειρο. Ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι η απάντηση, είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τους πολίτες. Προέρχεται από το παρελθόν και στο παρελθόν ανήκει. Δεν αποτελεί απάντηση για το μέλλον μας. Οπότε ναι, βεβαίως. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, την κρίση όμως, η κύρια απάντηση στην κρίση αυτή είναι να μάθουμε ε, τα μαθήματά μας και να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό όνειρο, όπως είπατε. Ε, για το άλλο ερώτημα δεν ε, θα αποφασίσω εγώ. Είπαμε ότι δεν θα, δεν θα είμαστε μια υπερφιλόδοξη προεδρία. Ίσως ο κύριος πάει να είναι πιο αρμόδιος να απαντήσει γι' αυτό. Η κυρία Ρούλε κι άλλος Γερμανός βουλευτής, Γερμανίδα, θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική προεδρία και εξ ονόματος της και Μπάρμπαρα Βάιλερ, γιατί κάνατε πολύ καλή αρχή και θα ενθουσιαστούμε αν συνεχίσετε όπως ε, η προκάτοχος, η προκάτοχή σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Ε, βέβαια, πολλές φορές ε, όλα μας τα όνειρα δεν μετατρέπονται σε νομοθεσία και κύριε Μάντερσε θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση πολλές φορές μεταξύ πολιτικών συμφερόντων και συμφερόντων των καταναλωτών. Δεν ταυτίζονται πάντα. Εμάς μας ενδιαφέρει να λάβουμε υπόψη μας τα τελευταία. Όχι κατά ανάγκη εκείνα των πολιτικών. Αυτό το λέω έτσι σαν ε, ε, μικρή παρατήρηση μετά από αυτά που είπατε. Κυρίως ήθελα όμως να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι έχετε μια ευκαιρία να ξεπαγώσετε αυτό το δύσκολο θέμα, να το προωθήσετε, γιατί είχαμε φτάσει σε αδιέξοδο. Ευχαριστούμε και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ήμουν σκιώδης, η Προεδρία σας κατάφερε πολλά και νομίζω ότι δεν απέχουμε πια από, πολύ από το να βρούμε συμβιβαστική λύση. Τώρα, δύο λόγια για την, ε, τους καταναλωτές και την εποπτεία της αγοράς. Είναι αξιοθαύμαστο ε, αυτό που κάνετε. Να προσθέσω όμως κάτι ακόμα, γιατί υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Πρέπει να πούμε κάτι. Εκ των προτέρων ήταν σαφές ότι η αρχή της χώρας προέλευσης θα δίχαζε το Συμβούλιο. Αυτό το ξέραμε από πριν. Επίσης ξέραμε ότι η εποπτεία αγοράς και η προστασία καταναλωτών δεν είχαν άμεση σχέση με το θέμα και χωρίς αυτό θα μπορούσε να λυθεί το θέμα. Ε, αλλά δεν προχώρησαν και δυστυχώς πήρατε τώρα αυτό το δώρο των αχαιών από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας, αλλά ε, δεν νομίζω ότι θα φταίτε εσείς αν δεν τα καταφέρουμε. I, Συμφωνώ μαζί σας κυρία Ρούλε. Και μάλλον, μάλλον στο μέλλον θα έρθω στο κόμμα σας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπατε, αλλά σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Μόζε θα συνεχίσει για την ασφάλεια των προϊόντων και ο κύριος Πουπάκης, ο κύριος Κοφεράτη, ο αντιπρόεδρος Κοφεράτη, ε, ο κύριος Κρυαντεκάμπος, ο κύριος Αγναλούγας, ο κύριος Σάριας. Άλλος. Θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, τώρα θα, πάρουμε, θα σας πάρουμε τους ομιλητές κατά δύο. Και να συνοψίσει μετά. Ε, η κυρία Σάλτε Μόζερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να έρχεστε εδώ και να ε, περνάτε το μήνυμα ότι δεν καταφέρατε σήμερα να, έχετε, να πάρετε εντολή. Εγώ όμως πρέπει πρώτα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας. Ξέρω ότι εργαστήκατε σκληρά για μια διαπραγματευτική εντολή. Όπως και η κυρία Ρούλε, πιστεύω και εγώ ότι δεν είναι ευθύνη της ελληνικής προεδρίας ότι δεν τα καταφέρατε. Έχω δει τις προτάσεις, καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο δεν θα δεχτεί την εντολή διαπραγματεύσεων γιατί η εντολή δεν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Εμεί έχουμε ένα σαφές μήνυμα, μια σαφή ε, άποψη για το... Εμείς αποστήλαμε το μήνυμα σχετικά με το Made in, όπου υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Είπαμε όμως ότι είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πω ότι τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα με τις χρονικές πιέσεις που τόσα προβλήματα δημιουργούν. Αν δεν εξευρεθεί λύση αύριο, δεν έχουμε εναλλακτική. Δεν υπάρχει δηλαδή, χάνεται η ευκαιρία για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, όχι εσάς, την Ελληνική Προεδρία, το Συμβούλιο. Θα κοιτάξουμε να πάμε την έκθεση στην Ολομέλεια και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Πρέπει όμως να πω επίσης και το υπογραμμίζω ότι δεν φταίει η ελληνική προεδρία, αλλά πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από το Συμβούλιο και το πώς δρά στο θέμα αυτό το Συμβούλιο. Όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε πιο λειτουργική εσωτερική αγορά. Όλοι ήταν ευτυχεί σε σχέση με την πράξη 1 και 2 για την ενιαία αγορά. Και τώρα έχουμε στο τραπέζι προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και ποιος είναι κατά, το Συμβούλιο ε, είναι κατά. Διότι αφού δεν θέλει να δώσει εντολή, αυτό σημαίνει στην πράξη ότι είναι κατά και δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αυτό είναι πρόβλημα πραγματικό. Εμείς τώρα είμαστε σε προεκλογική φάση και μιλώ με πολύ κόσμο. Πολλές φορές ε, με ρωτούν γιατί δεν έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, πιο δίκαιη ε, εσωτερική αγορά. Και τους λέω, ρωτήστε το Συμβούλιο γιατί αυτοί φταίνε. Και όταν οι καταναλωτές με ρωτούν γιατί έχουμε ακόμα επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά, τότε τους απαντώ πάλι το Συμβούλιο φταίει. Αυτό δεν κάνει αυτό που πρέπει. Είμαι λίγο ξεκομμένη και ομής. Ε, είναι κρίμα. Όμως ξέρω ότι προσπαθήσατε πραγματικά και... Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα γίνεται τίποτα άλλο. Θα πάμε στην Ολομέλεια και μετά θα πάμε στην προεκλογική εκστρατεία λέγοντας τι θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο. Γιατί εξακολουθεί να ισχύει το αίτημα για καλύτερη αποπτία της αγοράς και ασφαλέστερα προϊόντα. Άκουσα όμως ε, αυτό που είπατε αν έχουμε καλές ιδέες. Έχουμε καλές ιδέες. Ε, απόψε έχουμε μια συνάντηση Ήδη το ξανασυζητήσαμε το θέμα και πρέπει να σας πω νομίζω ότι μια από τις λύσεις θα μπορούσε να ήταν να δούμε τι κάνουν οι Αμερικανοί με το Made in. Εμείς ε, είχαμε διαπραγματεύσει με τις Ηνωμένες για τις εμπορικές συμφωνίες. Είπα αυτό το Made in το έχουν για τα εισαγόμενα αγαθά. Θα μπορούσαμε να το αντιγράψουμε να δούμε ποια νομοθεσία έχουν, γιατί ήδη πολλοί κάνουν εξαγωγές στη ΣΥΠΑ. Και αν ακολουθούσαμε την νομοθεσία τους, τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και να μην υπάρχει πρόβλημα. Είναι τρόπος αυτός για να λύσουμε το πρόβλημα του άρθρου 7. Εξακολουθώ να πιστεύω. Λοιπόν, και πάλι ξέρω ότι εσείς προσπαθήσατε. Ξέρω επίση ότι θα μεταφέρετε το μήνυμα σε όλο το Συμβούλιο ότι είμαστε ιδιαιτέρως απογοητευμένοι εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που θα αντιμετωπίσουμε τους πολίτες τους επόμενους μήνες, όχι το Συμβούλιο. Ξέρουμε δηλαδή ποιον θα κατηγορήσουμε. Λοιπόν, εμείς τώρα, ε, μπορεί να, μακάρι να βρεθεί λύση αύριο μεθαύριο, αλλά κατά τα άλλα πάμε για ολομέλεια. Ο κύριος Πουπάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, φίλε Κώστα, θα ήθελα να σα απασχολήσω με τη νέα σου ιδιότητα και εκτός Ελλάδος. Και θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Η κοινή έκθεση για την απασχόληση που συνοδεύει την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη αναφέρει πως σε κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα η μείωση του εργασιακού κόστου και η συγκράτηση των μισθών συνέβαλαν με αργού μισθού στην εξέλιξη των τιμών, ενώ παράλληλα η αύξηση των έμεσων και άμεσων φόρων μείωσε κατά πολύ το ποσοστό του διαθεσίμου εισοδήματο. Πράγματι, παρά την οικονομική ύφεση και τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητα που έχουν προκαλέσει μεγάλη πτώση τη κατανοητική ζήτηση και οι τιμέ στην αγορά εξακολουθούν να παραμένουν στα ύψη. Μάλιστα, σε πολλέ περιπτώσει οι τιμέ στην Ελλάδα στα είδη πρώτη ανάγκη εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένε σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, λαμβάνοντα υπόψη ότι 9 στου 10 Έλληνε καταναλωτέ έχουν αλλάξει τι καταναλωτικέ του συνήθειε, ενώ 4 στου 10 δυνατόν να αγοράσουν τα απαραίτητα είδη πρώτη ανάγκη. Θα ήθελα λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, σε ποια συγκεκριμένα μέτρα πολιτική αποτελεσματικέ δράσει σκοπεύετε πιθανόν να προβείτε σαν Προεδρία για τον εξορθολογισμό και την άμεση αποκλιμάκωσης των τιμών με στόχο την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την αποκατάσταση της καταναλωνικής δαπάνης. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Σαλτεμόζε, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να δώσουμε στο διάλογο μια ευκαιρία. Δεν λέω να έχουμε διάλογο αέναο χωρίς ε, λόγο και χωρίς ουσία, αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο, ε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την σύντομη χρονική περίοδο της μίας εβδομάδας δέκα ημερών για να προσπαθήσω να βρω μία λύση. Και είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε κάθε πρόταση και την πρόταση στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Δεν λέω ότι θα την εγκρίνουμε γιατί πρέπει πρώτα να την εξετάσουμε. Αλλά βεβαίως θα περάσουμε το μήνυμα στην μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Ακόμη και κατά το Σαββατοκύριακο είμαι στη διάθεσή σας. Όποια στιγμή θέλετε. Επτά μέρες την εβδομάδα δουλεύουμε στην Ελλάδα μετά την κρίση. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους προβλήματα διαθεσιμότητας. Μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά για να βρούμε μια λύση. Γιατί όπως ορθώς είπατε, θα ήταν κρίμα μετά από αυτή τη συζήτηση σε επίπεδο κοινοβουλίου, σε επίπεδο συμβουλίου, μετά από τόση πρόοδο, τελικά να μην υπάρχει συμφωνία λόγω του προβλήματος ε, Made in και της σχετικής ρήτρα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την εξέβρεση λύσεως, για να συμφωνήσουμε. Μιλήσω ελληνικά. Ε, αναφέρθηκε στην προστασία των καταναλωτών αυτό εδώ το Κοινοβούλιο πάντοτε είχε ευαισθησία για την προστασία των καταναλωτών, γι' αυτό και τούτη εδώ Επιτροπή, θυμάμαι όταν συναστήθη, δεν ονομάστηκε Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, αλλά Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Το θέμα αυτό είναι κομβική σημασία στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο γιατί έχουμε την ε, μεγάλη οικονομική κρίση η οποία μείωσε τους μισθούς και αύξησε δραματικά την ανεργία. Οι τιμές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί, αλλά όχι τόσο πολύ όσο έχουν μειωθεί οι μισθοί. Σε αυτό πρέπει να είμαστε καθαροί. Σε σχέση με το μέσο όρο των ε, ε, τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2011 εμείς είχαμε το 95%, το 2012 το 90%, το 2013 το 85%. Οι μισθοί όμως είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτό το επίπεδο. Επομένως χρειάζεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Η ύφεση είχε εκ των πραγμάτων ένα αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των ε, ε, τιμών διότι περιορίστηκε η ζήτηση και λειτουργήσαν σε ένα βαθμό οι νόμοι της ε, ζήτησης και της προσφοράς. από την άλλη πλευρά και σε κυβερνητικό επίπεδο ελήφθησαν διάφορα μέτρα χαρακτηριστικά θέλω να πω τις καινούργιες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν σε περισσότερες εταιρείες να πολλούν περισσότερα προϊόντα σε περισσότερα σημεία, αντιμετωπίζοντας δισκαμψίες στην αγορά και, και έτσι ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. Επίσης, ε, υιοθετήσαμε ένα καινούριο πλαίσιο για τη λειτουργία των καταστημάτων και της αγοράς, το οποίο μεταξύ των άλλων προβλέπει και μια απελευθέρωση σε σχέση με τις εκτόσεις, τις προσφορές και διεύρυνση των εκπτωτικών περιόδων ακριβώς για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για χαμηλότερες τιμές. Και τώρα, σε συνεργασία με τον ΟΣΑ και αφού μελετήθηκε το θέμα επί ένα χρόνο, προγραμματίζουμε μια μεγάλη οριζόντια παρέμβαση η οποία θα, αναφέρεται, θα αφορά σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς όπου έχουμε μια υπερπροστασία ορισμένων κοινωνικών ομάδων οι οποίες ε, κερδίζουν ε, ε, στην πραγματικότητα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και εις βάρος των, των καταναλωτών. Καταλαβαίνω είναι, είναι εύλογο εκείνες οι κοινωνικές ομάδες να υπερασπίζουν τη θέση τους, καθένας θα το έκανε, αλλά από την άλλη πλευρά είναι εξίσου εύλογο και η κυβέρνηση μέσω των, της προσπάθειας να αρθούν αυτά τα barriers του entry, τα, τα εμπόδια εισόδου στην, στην, στην, αγορά και μέσω της αποκατάστασης των κανόνων ανταγωνισμού είναι εύλογο η κυβέρνηση να επιδιώκει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό σε μια σειρά από κομβικούς τομείς της ελληνικής αγοράς θα επιδιωχθεί να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να έχουμε ε, το αποτέλεσμα που πρέπει. Άλλωστε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που κάναμε, μικρή λεπτομέρεια ίσω, αλλά είναι ενδεικτικό, αυτό που έγινε με το βρεφικό γάλα, που από τότε που επετράπη να μην είναι μόνο στα φαρμακεία αλλά και στα σούπερ μάρκετ, έπεσαν οι τιμέ κατά 20%. Ε, όλες οι μελέτες δείχνουν ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι αυτό που μετράει τελικά είναι ο καταναλωτής και κυρίως ο φτωχός άνθρωπος, αυτός που έχει πληγεί από την κρίση ο εργαζόμενος που είδε το εισόδημά του να περιορίζεται και ακόμη περισσότερο φυσικά ο άνεργο που συντηρείται από κοινωνικά επιδόματα ή από την οικογένειά του. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος ο κ. Κονφεράτη και ο καθηγητής ο κ. Δεκάμπος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί θέλουμε να μας τελειώσει ο χρόνος. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Υπενθυμίσατε στην παρουσίασή σας, στην εισαγωγή σας, το ότι η ελληνική προεδρία επηρεάζεται από αυτή την ε, ανώμαλη διάρκεια, την ανώμαλη περίοδο. Δηλαδή η Προεδρία είναι πιο σύντομη από ό,τι είναι για τις άλλες χώρες. Αυτό προφανές, προφανώς είναι ένα όριο, αλλά μπορεί να είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία. Διότι δικαιολογεί το ότι μπορείτε να επικεντρωθείτε επί λίγων νομοθετημάτων που έχουν όμως χαρακτήρα προφανώς και συμβολικό της Ευρώπης. Δείχνουν την Ευρώπη που θέλετε να προωθήσετε για το, να δημιουργήσετε στο μέλλον και να προωθήσετε. Κάποια θέματα από αυτά ήδη συζητήθηκαν από ε, αυτή τη ευκαιρία έχουν ανάμεσά τους βάρος και αξία διαφορετική. Θα ήταν σοβαρός περιορισμός εάν όπως αναφέρθηκε από, πριν από λίγα λεπτά, η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων δεν φτάσει στο λιμάνι τελικά. Θα ήταν ένα σήμα απαραίτησης προς τους ε, καταναλωτές και τη μελλοντική Ευρώπη που θέλουμε. Ε, πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό θα ήταν αν αντίθετα φτάσουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επιληθεί και το θέμα της ασφαλείας των προϊόντων. Θα ήταν σημαντικό αν φτάσουμε σε θετικό, σε θετική κατάληξη όπως ευχηθήκατε εσείς και έχετε και πρόθεση να προσπαθήσετε να πετύχετε, να εντοπίσετε λύσεις που επιτρέπουν να έχουμε πόρους πρόσθετους που μπορούμε να δεθέσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις εργασίες αυτέ της ε, Επιτροπής μας θα δείτε αναφορά στις οδηγίες που συζητούνται ακριβώς πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα σημαντικό, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για αύριο. Διότι δεν είναι μια ε, υπόθεση, δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη σε αυτό το κόσμο αν δεν έχουμε, αντιμετωπίσουμε και το θέμα της όρευσης μέσω της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια και στη σύντομη αυτή διάρκεια έχετε και δικαιολογία πολιτική για να το στηρίξετε αυτό και να το επιδιώξετε αυτό. Ευχαριστώ. κύριος Κάμπος. Thank you, Chair. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπουργέ, καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι σας. Έχω να πω κουβέντες αλληλεγγύης για σας, γιατί και στη χώρα μου υποφέρουμε από τα ίδια προβλήματα όπως και στη δική σας. Ε, ίσως είμαστε πιο ευχαριστημένοι τις δύο τελευταίες εβδομάδες διότι από ό,τι φαίνεται οι αγορές αρχίζουν να υπόσχονται κάποια πράγματα για όλες τις χώρες μας. Αυτό είναι παράξενο. Δεν υπάρχει διάκριση. Και γνωρίζουμε ότι η καλύτερη απάντηση στην οικονομική ύφεση, μία καλή απάντηση είναι η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση των κοινών αγορών για ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες και βελτίωση της έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας. Κάτι που αναφέρατε, συμμερίζομαι τις προτεραιότητες σας απόλυτα όσον αφορά την τεχνική τυποποίηση, να αναπτυχθεί το θέμα των ταξιδιών, των πακέτων ταξιδιών, θα είναι κάτι πολύ θετικό όπως για χώρες όπως είναι οι χώρες μας και υποπτία της αγοράς, ηλεκτρονική τιμολόγηση και καταπολέμηση της ε, κατάκτησης αγοράς από ομιλού συμφερόντων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είχαμε τις βρεφικές τροφές. Ε, είχαμε παραδείγματα από τις χώρες μας. Ας, αρπάξουμε, ας αδράξουμε την ευκαιρία για να ε, καταπολεμήσουμε αυτή την κατάκτηση αγοράς στους μεγάλους ομίλους να σας υπενθυμίσω κάτι που γνωρίζετε. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η χθεσινή, για την παγκόσμια οικονομία, περιέχει βασική λέξη στις συστάσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δύο λέξεις κλειδιά περιέχονται. Στοχευμένη δανειοδότηση, target lending, στοχευμένη δανειοδότηση. Αυτό που ανέφερε ο Σέρτζιο Κονφεράτη, δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε και εδώ. Εμείς στην Ευρώπη δεν εφαρμόζουμε μέτρα ε, ποσοτικής διευκόλυνσης και ελαστικοποίησης, τότε ας επιβάλλουμε την στοχευμένη δανειοδότηση, αφού δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι ΙΠΑ. Και έτσι πιστεύω ότι θα μπορούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ευχαριστώ. There Υπήρξε κάτι κοινό στις δύο τελευταίες παρεμβάσεις. Η προστασία των καταναλωτών, η διάσταση της προστασίας των καταναλωτών. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το πακέτο για τους καταναλωτές, ας το πούμε έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Διότι θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό σε αυτή τη φάση να μην διεκπαιρεωθεί το θέμα αυτό. Θα ήταν πολύ αρνητικό για τους καταναλωτές και θετικό μόνο για τους ευρωσκεπτικιστές και τον ευρωσκεπτικισμό. Μόνο οι ευρωσκεπτικιστές θα κερδίσουν εάν αποτύχουμε εμείς, αν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Διότι δεν είναι ένα τεχνικό πακέτο, δεν είναι κάτι περιττό, δεν είναι κάτι δευτερεύουσα σημασίας, είναι κάτι σημαντικό, κατανοητό από τους πολίτες, κατανοητό από τους ε, καταναλωτές. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να πολεμάμε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία και είμαι βέβαιος ότι όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή ότι ο καταναλωτής θα είναι στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας, πρέπει να προστατευτεί. Σε κάποιες χώρες οι οργανώσεις καταναλωτών δεν είναι πολύ ισχυρές, αλλά εξαρτάται από τους θεσμούς να προστατεύσουν τους καταναλωτές διότι εκείνοι που είναι καλά οργανωμένοι, τα διάφορα λόμπι, οι ομάδες πίεσης έχουν τη δύναμη να ασκήσουν πίεση επί των κυβερνήσεων, επί των κοινοβουλίων, ούτως ώστε να ενισχύσουν τη δική τους θέση ή να διατηρήσουν τα προνόμια τους. Κάποιος όμως πρέπει να φροντίσει τον καταναλωτή. Αυτή είναι η πεποίθησή μας, αυτή είναι η αρχή μας και είναι ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του εξαμήνου, του εξαμήνου της ελληνικής ε, προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στην καρδιά μας ε, την προστασία του καταναλωτού στο επίκεντρο των εργασιών μας. Λοιπόν, τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Να είσαστε φιδωλίους όσον αφορά το χρόνο, συνάδελφοι, να έχουμε χρόνο για απαντήσει. Η κυρία Σενέλοβα, ο κύριος Αρίας και ο κύριος Ταραμπέλα. Τον άφησα, ήμουν ανεκτικό και τον άφησα κάπω να παρισφρήσει, αλλά ήταν συγγητή μα και έχει να αντιμετωπίσει περισσότερε τροπολογίε από ό,τι όλοι οι υπόλοιπα, υπόλοιποι τα τελευταία τρία χρόνια. Και κυρία Ντανιέλ, η άλλη αντιπρόεδρο. Θα σα ακούσουμε πρώτα. Λοιπόν, Όλγα. Θα μιλήσω τσεχικά, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ε, Vážený ε, Αξιότιμε κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ως εισηγήτρια ασχολήθηκα με το σύστημα e-call, τις ηλεκτρονικές κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Ε, βέβαια, ε, στην αρχή φοβήθηκα ότι δεν θα μιλούσατε καθόλου για το e-call. Μετά όμως το θίξατε είναι ένα από τα θέματα για τα οποία θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική προεδρία, διότι εκείνη, όπως και το Κοινοβούλιο, θεωρεί το νομοθέτημα αυτό πολύ σημαντικό, γιατί ο σκοπός είναι να μειωθούν ε, οι θάνατοι από τα τροχαία. Ε, και εσείς αναφέρατε το όφελός του για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δουλεύουμε ε, για εδώ και καιρό το θέμα. Δεν είναι καινούριο. Για το e-call μιλάμε εδώ και δέκα χρόνια. Πολύ εντατικά και πολύ εντατικά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είμαστε στην τελική ευθεία και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας το Φεβρουάριο. Είπατε ότι θα δούμε πόσο θα προχωρήσει το θέμα. Καλό θα ήταν να έχετε τη φιλοδοξία να καταλήξετε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να φτάσετε μέχρι εκεί. Και εγώ ως εισηγήτρια ε, χαίρομαι που θα συνεργαστούμε εντατικά. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Άριας Ετσεβερία. Mm. Σας καλωσορίζω ως πρώην Ευρωβουλευτή και νυν Υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αυτό αποδεικνύει το έργο της ελληνικής κυβέρνησης και το ενδιαφέρον της για το ευρωπαϊκό πνεύμα. Προφανώς ο ευρωσκεπτικισμός καλπάζει και στη χώρα σας και αλλού στην Ευρώπη. Εγώ όμως σας καλωσορίζω, αρχίσατε να μιλάτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο σημαντικές για την απασχόληση και τη μεγέθυνση και την οικονομία. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, ε, γιατί τρέχει ο χρόνος. Καταρχήν να υπογραμμίσω το θέμα αυτό του Made in Μιλήσαμε για έξυπνες λύσεις. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε προς την εξέβρεση λύσης, συμφωνίας ε, που θα είναι υπέρ της ε, ε, ενίας αγοράς, που θα καταργεί τα εμπόδια που υπάρχουν. Νομίζω ότι το made in είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας μπορούν έτσι να ε, βελτιώσουν το δυναμικό τους και είναι και σημαντικό ως ενημέρωση για τους καταναλωτές που θα γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων, τα ε, ευρωπαϊκά προϊόντα κλπ. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η ελληνική προεδρία πρέπει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ασφάλειας των προϊόντων και της προστασίας των καταναλωτών. Αυτός είναι ένας στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, συνθήκης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, γιατί και αυτό έχει να κάνει με την απασχόληση και την ανάπτυξη. αυτό το θέμα δεν είναι μόνο στην Ισπανική ημερήσια διάταξη αλλά και στην Ευρωπαϊκή. Κυρίως αναφέρομαι εδώ στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Μπορείτε να σκεγγραφίσετε κάποια λύση εδώ ή να αναφέρετε κάποιες, εθνικ... Ε, κάποιες ε, ε, θετικές εξελίξεις. Κύριο Σταραμπέλα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω, γιατί έχουμε και την οδηγία της απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αν θυμάμαι καλά, είχατε κι εσείς γνωμοδοτήσει ε, για αυτήν την ε, έκθεση το 2006. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση που θα σας κάνω, γιατί σε σχέση με τον ε, πολίτη, τον καταναλωτή, μιλήσατε και για τους άνεργους, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να δω να γεννιέται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, να υπάρχει απελευθέρωση αλλά και το αποτέλεσμα αυτών. Γιατί μιλάμε για ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές, είμαστε στο τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πρόθεση απελευθέρωσης πάρα πολλών τομέων και υπηρεσιών να κάνουμε ένα check-up, έναν έναν έλεγχο του κατά πόσο έχει υπάρξει πρόοδος, πού έχουμε κάνει τις περισσότερες ε, πρόοδους και τις λιγότερες πρόοδους. Ε, από απόψεως αποτελεσματικότητας υπηρεσιών προς τον ε, πολίτη, είναι λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικές για τον πολίτη. Το κόστος στοιχίζει λιγότερο η ενέργεια σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Όπως επίσης και το επίπεδο της ποιότητας των, της απασχόλησης στην παροχή υπηρεσιών. Το επίπεδο ε, των μισθών για παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν ίσως θα έπρεπε να τα συνυπολογίσουμε ε, να, προσθέσουμε να, να συγκρίνουμε ε, και τις αστικές περιοχές με, τις, με την Ήπεθρο ε, γιατί πολλές φορές ε, η Ήπεθρος έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα να πληρώσει σοβαρό τίμημα ε, σε σχέση με τις αστικές περιοχές και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε, αν θα ήταν χρήσιμο όχι μόνο ενημερωτικός αλλά και ως γνώμονα για το μέλλον να έχουμε έναν πραγματικό έλεγχο των διαφόρων απελευθερώσεων που έχουν γίνει ως τώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Η κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας καλωσορίσω, να σας ε, ευχηθώ καλή τύχη και καλό κουράγιο, γιατί δεν είναι απλή η κατάσταση. Έχετε μια πολύ σύντομη προεδρία μπροστά σας, αλλά και πολύ σύντομη θα πει, όπως είπε και ο κύριος Κοφεράτη, ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία. Οπότε θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας. Μιλήσατε για την απασχόληση και για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλήσατε για την έρευνα και την καινοτομία. Ξέρετε ότι στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο πολλές φορές μετά από πολλές συζητήσεις ε, για τον προϋπολογισμό και στην Επιτροπή μας ε, ασχοληθήκαμε με θέματα κλειδιά για τη βελτίωση της απασχόλησης, της συνεργασίας ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Επίσης προσθέσαμε 30% στον προϋπολογισμό τον ερευνητικό. Έρευνα και καινοτομία είναι το κλειδί της ανταγωνιστικότητας και της ε, απασχόλησης. Και το λέω αυτό γιατί το βλέπουμε και στις χώρες μας και στις μικρές μας περιφέρειες. Βλέπουμε συχνά ότι η έρευνα ε, οι ερευνητές δουλεύουν στη γονίτσα τους και δίπλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και εκείνες λίγο απομονωμένες μήπως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς μπορούμε παντού να έχουμε ε, εσωτερική αγορά ομοιόμορφα, αν υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ε, δικτύων και σε εθνικό επίπεδο αλλά και δρασυνοριακά, ε, μέσω για παράδειγμα διαφόρων ε, ε, γραφείων που να μειώνουν την γραφειοκρατία για παράδειγμα. Προς όφελος όλων και των Ευρωπαίων πολιτών κυρίως βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κι εγώ κάτι γιατί πήγαμε στο ψηφιακό κέντρο καινοτομία στην Αθήνα και εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ. Ε, ίσως ε, θα μπορούσατε να μας πείτε και ορισμένα πράγματα για το πόσο καλά πηγαίνουμε ως προς τα θέματα της, της καινοτομίας. Λοιπόν, κυρία Σενιλόβα, ε, <laughs> okay. Ε, πράγματι το e-call ε, no, I, ε, I have to speak Greek, English, English, okay. Uh, indeed. Ας τα πω στα αγγλικά. Η οδηγία e-call είναι πολύ σημαντική οδηγία. Έχουμε να διχειριστούμε κατεπηγόντως. Δεν είμαι υπεύθυνο όμως εγώ, το είπα. Είναι υπεύθυνο ο υπουργό ε, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών. Εκείνο το χειρίζεται. Είναι σημαντικό για τους πολίτες, για την οδική ασφάλεια. Σημαντικό για να αποφεύγουμε θύματα από τροχέα. Και στις μεσογειακές χώρες είναι περισσότερα τα θύματα ε, στους δρόμους από ότι σε άλλες χώρες. Οπότε πρόκειται για εθνική προτεραιότητα μεταξύ άλλων. Όπως είπα, θα προχωρήσουμε το θέμα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Οι προβλέψεις από τις υπηρεσίες μας είναι ότι δεν επαρκεί ο χρόνος για να κλείσει ο φάκελος. Γι' αυτό είπα ότι θα τελειώσει η πρώτη ανάγνωση και η δεύτερη θα γίνει επί Ιταλικής Προεδρίας. Βέβαια, αν υπάρξουν εξελίξεις, ταχύτερα από ό,τι περιμένουμε, τόσο το καλύτερο. Θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσετε και θα γίνουν συζητήσεις και στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Αλλά μόλις ε, το πιάσαμε το θέμα, δεν ήταν ένας φάκελος όπου οι Λιθουανοί είχαν προχωρήσει, δεν το είχαν πιάσει, λόγω χρονικών περιορισμών. Δεν θέλω δηλαδή να κατηγορήσω κανέναν εδώ. Έτσι έχει το πράγμα. Κύριε Αριάς, μιλήσατε για την κρίση. Εμείς είμαστε τα θύματα της κρίσης. Και η δική σας η χώρα και η Πορτογαλία, αναμφιβόλως. Εμείς έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την κρίση. Μέχρι τώρα καταφέραμε να έχουμε κάποια ορατή πρόοδο σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή. Έχουμε το πέμπτο χαμηλότερο έλλειμμα σε όλη την Ευρωζώνη τώρα και έχουμε παρά τις προβλέψεις έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι ανεμένετο. Υπάρχει στον προϋπολογισμό μας πρωτογενές πλεόνασμα και σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ για την ανάπτυξη, η μεγέθυνση, η Ελλάδα είναι πρωταθλητής ανάμεσα στις χώρες του ΩΣΑ στις διαφορετικές αλλαγές τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα και δεν μπορούμε έτσι να κεφαλαιοποιήσουμε την πρόοδο. Ως ένα βαθμό αυτό ισχύει και για τη δική σας χώρα και για άλλες χώρες. Ε, ένα πρόβλημα είναι η ρευστότητα, το πρόβλημα με τη ρευστότητα και ο τραπεζικό τομέα. Η ρευστότητα πλήττει τη μιμία. Και αυτός ο κρίκος που λείπει συνδέεται με έναν άλλο παράγοντα που είναι η εμπιστοσύνη, ο παράγον εμπιστοσύνη. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για το στόχο της ε, δημοσιονομικής ε, προσαρμογής και την ε, υιοθέτηση νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά μας. Παράλληλα, νομίζω ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράσει με πιο ορατό τρόπο την αλληλεγγύη της με τις χώρες μας. Δεν υποτιμώ την ε, βοήθεια καθόλου, αλλά όλες οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κρίσιμη καμπή και πρέπει τώρα να δώσουμε μια νέα όθηση στις προσπάθειες, ούτω ώστε, όπως είπατε πολύ σωστά, να μειωθεί η ανεργία κυρίως των νέων. Βεβαίως έχουμε την εγγύηση για την νεολαία, έχουμε τους νέους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν επαρκούν. Πρέπει να αναζωογονήσουμε τις οικονομίες μας. Και βέβαια έχουμε μια βάση για να στηριχθούμε, έναν πυλώνα αν θέλετε, που είναι η δημοσιονομική η πρόοδος στη δημοσιονομική προσαρμογή και η πρόοδος στην ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πρέπει να ε, λύσουμε και τα άλλα θέματα, τα άλλα προβλήματα, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα και την εμπιστοσύνη, τον παράγοντα εμπιστοσύνη. Έτσι ερμηνεύω εγώ την κατάσταση και σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά τις χώρες μας, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε, όχι γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε προς κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αλλά γιατί είναι πατριωτικό καθήκον μας. γι' αυτό είναι τόσο απλό. Οι λαϊκιστές πάντα μιλάνε για εύκολες λύσεις και ε, ε, ε, δείχνουν στον κόσμο μαγικές λύσεις. Αλλά αυτές δεν είναι λύσεις, είναι ένα πρόβλημα ακόμα όλο αυτό. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό τον ρεαλιστικό, πραγματιστικό τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης. Ε, κύριε Ταραμπέλα, η απελευθέρωση δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η ενιαία αγορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, όπου έχουν απελευθερωθεί τα πάντα και υπάρχουν και χώρες όπως η Γαλλία για παράδειγμα, όπου υπάρχουν και κάποιες κρατικές παρεμβάσεις. Εξαρτάται από το κράτος μέλος. Ε, στο κράτος μέλος εναπόκειται να πάρει τις αποφάσεις εδώ η, η απόφαση του 87 την ενία πράξη του Λουξεμβούργου και το 1992 μετά για την ενία αγορά, αφορούσε τη δημιουργία ενιαίας αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να είμαστε ανταγωνιστικοί στην ενία αγορά πρέπει η κάθε χώρα να λαμβάνει σε εθνικό επίπεδο τις αποφάσεις της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συμμορφούνται όλοι προς τους κανόνες του παιχνιδιού και ε, το βασικό εδώ είναι η ενιαία αγορά. Αυτή η προσέγγιση υιοθετήθηκε για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κυρία Βερνιό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σχετικά με την, ε, τις δυνατότητες που έχουν οι ευρωπαϊκές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να εστιάσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και στο, να εστιάσουμε επίσης και στον παράγοντα της καινοτομίας. Σήμερα πήγα στην Επιτροπή Ήτρε και τους μίλησα για την ε, βιομηχανική πολιτική και είπα ότι έχουμε πέντε αρχές ή πέντε πυλώνες στην προσέγγιση μας, ε, στην προσέγγιση της Προεδρίας μας, που είναι η καινοτομία, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η μείωση του ενεργειακού κόστους και δύο ακόμα που δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Η μείωση της γραφειοκρατίας που είναι ουσιώδες θέμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το στόχο ε, καταργώντας την ε, περισσή γραφειοκρατία και η επικέντρωση στις δεξιότητες για να ενισχύσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Πρέπει να συνδυάσουμε κάποιες ε, συγκεκριμένες παραμέτρους Επαναλαμβάνω όμως ότι η στήριξη της βιομηχανίας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κοινωνική πολιτική, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να διασώσουμε θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε νέες. Γι' αυτό ήταν σοβαρό λάθος της Ευρώπης που παραμέλησε τη βιομηχανική πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες. Εγώ τότε ήμουν Ευρωβουλευτής και θυμάμαι πολλές συζητήσεις για την περιβαλλοντική διάσταση ναι, που ήταν θετική και πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στο περιβάλλον, αλλά από την άλλη υποτιμήσαμε το ρόλο της βιομηχανίας και γι' αυτό είχαμε αρνητικές εξελίξεις. Τώρα η ΕΠΑ, η Κίνα έχουν θετικά ποσοστά μεγέθυνσης και η Ευρώπη είτε πλήττεται από ύφεση ή έχει πολύ μικρά θετικά ε, ποσοστά μεγέθυνσης. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στη βιομηχανία μας. Όχι επενδύοντα χρήμα κατά ανάγκη, αλλά μειώνοντα τη γραφειοκρατία, μειώνοντα το ενεργειακό κόστο, ε, ακολουθώντας τις πιο έξυπνες πολιτικές. Αυτή είναι μια προτεραιότητά μας. Δεν πιστεύουμε ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα επί ελληνικής προεδρίας, αλλά με βάση την ανακοίνωση για τη βιομηχανία της Κομισιόν, με βάση τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου, που η έκθεση Ράιζε που εγκρίθηκε το Δεκέμβρη πριν λίγο, ε, θα προσπαθήσουμε να ε, επιτύχουμε κάποια πρόοδο ώστε να δημιουργήσω μια καινούρια στέρεη βάση για να αναπτυχθεί η βιομηχανία μας. Αυτή την προσέγγιση έχουμε προκρίνει. Ευχαριστώ πολύ και πάντα είμαι στη διάθεσή σας να έρχομαι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να οργανώνουμε άτυπες συνεδριάσεις και σε τελευταία ανάλυση να λύνουμε προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Κύριε Υπουργέ Κώστα, μεγάλη χαρά μας που σε δεχτήκαμε εδώ συνεδρίαση. Ευχαριστώ που απάντησε τους πολλές ερωτήσεις. Ευρύ φάσμα κάλυπταν οι ερωτήσεις, ευρύτατο. Και νομίζω ότι κατάλαβες ότι ε, έχουμε προθυμία να βοηθήσουμε στα καθήκοντά σου. Η εμπειρία σου εδώ στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση σε κάνουν ιδεώδη για τη θέση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας που καλύπτει τόσους πολλούς τομείς όπως έδειξε σήμερα. Ελπίζουμε να έχει σημαντικές επιτυχίες και αν καταφέρουμε να ξανακαλέσουμε πριν πάμε στις εκλογές θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Για την ώρα καλή τύχη, την καλύτερη τύχη και προσβλέπουμε στην πρόοδο και ευχαριστώ και την ομάδα σου. Μεγάλη χαρά που βλέπουμε την Άρτεμη. Περάσαμε το χρυσό πρωί μαζί, ετοιμάζοντας ε, συμβιβασμού. Ε, για, τις, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που ελπίζουμε θα προωθεί τελικά μεγάλη επιτυχία. Να πω απλώς ότι εδώ ολοκληρώσαμε τη δημόσια συνεδρίαση την απογευματινή. Στις παρατέταρτο θα γίνει συνεδρίαση των συντονιστών. Πέρασε σας για το κοινό. Ευχαριστούμε και γεια σας.